Αν κατάλαβα καλά, αυτή ήταν μια παρατήρηση σχετική με τα πρακτικά και τις προσωπικές δηλώσεις. Ήταν μια αναφορά στις ε, παρεμβάσεις σας τις προηγούμενες. Έχετε κάποια άλλα σχόλια να κάνετε για τα πρακτικά της 9 με 13 Σεπτεμβρίου. Γίνονται δεκτά. Κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές της Ουγγαρίας με ενημέρωσαν ότι ο κύριος Ζόλταν Μπαγκό Αντικαθιστά την κυρία Ένικε Κιωρή από την 1η Οκτωβρίου του 2010. Κύριε Μπάγκο, καλωσορίζες τον κύριο Μπάγκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας παρατηρήσω επίσης ότι σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναμένει την απόφαση ελέγει μετά που θα ακολουθήσει τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων του. Περνάω στο επόμενο θέμα. Η υπογραφή πράξεων σύμφωνα με την κανονική νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 74 το περιεχόμενο θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά της